Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και η ομάδα των Ελευθεριών και Δημοκρατών ε, έχουν δώσει προτάσεις διορισμών στις επιτροπές και αντιπροσωπείες που καταγράφονται στα πρακτικά της τρέχουσας συνόδου. Εάν δεν παρουσιαστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνόδου θα εγκριθούν αυτές οι ε, υποψηφιότητε. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι δυνάμει του άρθρου 70